σκήνια συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών τάφων στην Ταϊλάνδη. Δίνω το λόγο στους συντάκτες του σχεδίου της πρότασης ψηφίσματος. Ο κύριος Κοράου έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η είναι μια εθνοτική ε, μειονότητα που διώκεται πολύ περισσότερο από άλλες. Πρόκειται για ένα έρμα το οποίο θέλουν να πετάξουν όλα τα έθνη. Ο λαός αυτός διώκεται από τους βουδιστές της ε, Μιανμάρ και βεβαίως διέφυγαν δια θαλάσσης. Είναι μια κατάσταση παρόμοια με της Μεσογείου διέφυγαν από τον κόλπο της Βενγάλης προς την Ταϊλάνδη, η οποία δυστυχώς έχει βασανίσει αυτό το λαό που βρίσκεται στην όμορη περιοχή με τη Μαλαισία. Η Μαλαισία και η Ινδονησία υποδέχονται αυτούς τους πρόσφυγες και θέλουμε να αποστείλουμε ένα στεναρό μήνυμα προς την ε, τα Ιλάνδη και το Μιανμάρ για να αλλάξουν στάση έναντι αυτού του λαού και να τηρήσουν τα ελάχιστα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Λοχμπίλερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη Νότια Ταϊλάνδη υπάρχουν πολλά κρυφά στρατόπεδα στα οποία ε, γίνεται συγκέντρωση και βασανισμοί, αναγκαστική εργασία και αποκλεισμός ε, με, ε, και απαγωγή με απέτηση λίτρων από τις οικογένειες των κρατουμένων. Έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 30 μαζικοί τάφοι. Ε, υπάρχει λαθρεμπόριο ανθρώπων και γι' αυτό πρέπει να γίνεται πιο αυστηρός έλεγχος των ε, ροών των ε, προσφύγων. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε ότι πρόκειται για τους Ροχίνγκα από τη Μιανμάρ, από τον Μπαγκλαντές. 25.000 ήταν αυτοί οι οποίοι, οι οποίοι πέρασαν αυτούς τους δρόμους. 8.000 άνθρωποι επί μέρες και, μην, και εβδομάδες περνάνε από πολύ σκληρές συνθήκες διαδρομές για να μπορέσουν να ξεφύγουν, δεν τους προσφέρεται ούτε νερό και πρέπει να αντιληφθούμε ότι ήταν Ινδονήσιοι σε εκείνοι οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία διέσωσαν τους ε, πρόσφυγες αυτούς. Πρέπει να ληφθεί μια απόφαση πολιτική ώστε να διασώζονται οι άνθρωποι αυτοί που κινδυνεύει η ζωή τους. Απαιτούμε και απευθύνουμε έκκληση να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο ανθρώπων το πάζαρο αυτό και πρέπει να διαδραματίσουμε εμείς κεντρικό ρόλο. Η κατάσταση των Ροχίνγκα στη Μιανμάρ είναι ε, απεγνωσμένη. Πρέπει να αλλάξει στάση απέναντι στους Ροχίνγκας η κυβέρνηση, πρέπει να τους χορηγήσει την ηθαγένεια και πρέπει να αλλάξει στάση δραστικά απέναντι στις διακρίσεις και τις διώξεις η κυβέρνηση της Μιανμάρ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος και τώρα η κυρία Χαράνσοβα. Πρόεδρε, το πρόβλημα της μετανάστευσης στην Μεσόγειο δεν μπορούμε να το δούμε μεμονωμένα. Η κρίση των προσφύγων Ροχίνγκια μας υπενθυμίζει την υποχρέωση αυτή να αναλάβουμε δηλαδή μια συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος μετανάστευσης άντρες, γυναίκες και παιδιά που προσπαθούν να ξεφύγουν από την ε, εθνοτική βία στη Βυρμανία, ε, φτάνουν ε, σε συνθήκες άθλιες μέχρι τη θάλασσα για να χάσουν εκεί τη ζωή τους. Λυπούμε ιδιαίτερως για την κατάσταση στο Ροχίνγκια. Χρειάζεται να τους δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία από τους εμπόρους. Η προσωρινή προστασία ωστόσο δεν θα λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα ούτε στα στενά του Μάλακα, ούτε, στα, ούτε στην Μεσόγειο λύνεται το πρόβλημα της ε, μετανάστευσης. Ε, πρέπει να ε, πατάξουμε τους δουλεμπόρους που εκμεταλλεύονται τις ανάγκες και τις ελπίδες των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα της μετανάστευσης και να δώσουμε λύσεις. Η Βυρμανία πρέπει να αλλάξει την προσέγγιση της εναντί των μειονοτήτων και να αναγνωρίσει τους Ροχίνγκια ως ε, πολίτες της με όλα τα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσάρλς Τάνοκ έχει το λόγο. Πρόεδρε, τις τελευταίες εβδομάδες στην Ευρώπη συζητήσαμε πολύ τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εμείς ω προς τους δικούς μας, προς, μετανάστες στην Μεσόγειο και την ανάγκη να τους προσφερθεί υποστήριξη σε σχέση με διώξεις και οικονομικές καταστροφές στη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Η μουσουλμανική μειονότητα των Ροχίνγκια στη Βυρμανία τώρα δείχνει αντίστοιχες ε, εικόνες με αυτές που γνωρίζαμε στη Μεσόγειο και στην ε, Νοτιοανατολική Ασία. Η Ινδονησία όμως και η Μαλαισία φαίνεται να δέχθηκαν να υποδεχθούν προσωρινά 7.000 πρόσφυγες τι δε τελευταίες ώρες ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της Γκάμπια την ε, πρόθεσή του να χορηγήσει μόνιμο καθεστώς πρόσφυγα σε όλους τους πρόσφυγες Ροχίνγκια. Μακροπρόθεσμα ωστόσο το μόνο που μπορεί να γίνει σαν λύση θα είναι να με χρειάζεται οι άνθρωποι αυτοί να ε, ξεκινήσουν το δρομολόγιο αυτό, το τόσο επικίνδυνο δρομολόγιο. Πρέπει το ζήτημα των Ροχίνγκια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Το δε ε, κόμμα της αντιπολίτευσης της Aung San χαίρομαι πάρα πολύ που ε, ζήτησε ε, πρόσφατα να λυθεί το ζήτημα των Ροχίνγκια και να τους χορηγηθεί η ηθαγένεια, να τους αναγνωριστεί η ηθαγένεια. Πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα αυτό και μέσα από τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βοήθειες που χορηγεί. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Merci. Ευχαριστώ. Τις τελευταίες εβδομάδες αποκαλύφθηκαν με τους σωματικούς τάφους ε, ε, θλιβερές καταστάσεις ε, στην χώρα αυτή υπάρχει σωματεμπορία, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα λίτρα έχουν τραγική μοίρα. Υπάρχουν και πολλοί Μπαγκλαντεσιανοί, αλλά και κυρίως Ροχίνγκοι, οι οποίοι φεύγουν από τη Βερμανία και το διωγμό, αλλά κυνηγούνται πάλι. Το ΑΣΕΡ μιλάει για 25.000 άτομα τα οποία ε, φεύγουν. Πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στις ακτές ε, των ε, όμορων χωρών και 8.000 επίσης αναζητούν άλλο καταφυγή. Διεθνείς αρχές όμως όπως και σε άλλες περιπτώσεις ε, δεν είναι στο, στο ύψος των περιστάσεων. Πολύ λίγα χρήματα έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 300.000. Είναι αυτοί όμως οι άνθρωποι θύματα διακινητών, ε, ε, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να γίνουν σωστά, να τους υποδεχθούν σε χώρες όπου δεν θα κινδυνεύουν. Κύριος Λένερς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μα σοκάρουν οι αποκαλύψει αυτών των ομαδικών τάφων ε, στην Ταϊλάνδη. Οι πρόσφυγες Ροχίνγκια που δολοφονήθηκαν ή απλά τους άφησαν να πεθάνουν από την πείνα ή από ασθένειες η κυβέρνηση της πραγματικά καλείται να διεξαγάγει αμέσως ε, έρευνα αξιόπιστη και εντελεχή για αυτούς τους ομαδικούς τάφους. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να βρεθεί και μία λύση για την ανθρωπιστική κρίση στη θάλασσα όπου χιλιάδες πρόσφυγες ε, πραγματικά βρίσκονται στις ακτές χωρίς ε, να μπορούν να τους εξασφαλιστεί καμία αξιοπρεπής ε, συνθήκη διαβίωσης. Όλες οι χώρες της περιοχής πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους και να συμμετάσχουν ε, τουλάχιστον στη δέσκεψη κορυφής στην Μπαγκόκ στα τέλη Μαΐου. Θα πρέπει βέβαια να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες ρίζες του προβλήματος που είναι η συνεχής διωγμή και διακρίσεις ε, κατά των προσφύγων Ροχίνγκια στη Μιανμάρ. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει πολιτική. Πρέπει να κάνει πάντο δυνατό για να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων όσων κατοικούν στην επικράτεια τη χώρα τη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Γιώσεφ Βάιντεν Χόλτσερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το κεφάλαιο της ζωής στο Ροχίνγκια είναι ένα από τα πιο μελανά στην ιστορία Πρόκειται για τον πλέον διοκόμενο λαό, την πλέον διοκόμενη εθνοτική ομάδα. Χρειάζονται όλοι μας την υποστήριξη. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα σε όλη την περιοχή, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε τη λιδία μύθο, λίθο της ε, δημοκρατικής διαδικασίας στην ε, Μιανμάρ. Και βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η λιδία λίθος της ε, ανθρωπιάς μας. Μια λύση λοιπόν με ανθρωπιά, μια ανθρωπιστική λύση για τους Ροχίνγκια είναι η μόνη λύση η οποία μπορεί να δοθεί και μπορεί να δοθεί μόνο στην ίδια την περιοχή. Εκεί που βρίσκονται οι Ροχίνγκια ως εθνική ομάδα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τη δυνατότητα στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας επιπλέον να αναλάβουμε δράση και να στηρίξουμε τα γειτονικά κράτη, για τα οποία είμαστε και ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο, όπω ο παραδείγμα των Μπαγκλαντέ. Ευχαριστώ. Οι εκπρόσωποι τώρα των πολιτικών ομάδων. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριο Σόγκορ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και με την κρίση με τους μετανάστες στο, στη Μεσόγειο, θεωρούμε ότι η μαζική αυτή έξοδος από το ε, Μιανμάρ δεν είναι κάτι το νέο. Το 2009 είχαν διασωθεί πολλοί ροχίνγκια αφού προσέφυγαν στη θάλασσα. Υπάρχει φτώχεια, βία και μεγάλος διωγμός. Τα πιο, ευάλωτε, πιο, οι πιο ευάλωτες ε, ομάδες επλήγησαν και αυτό το βλέπουμε και από τους ομαδικούς τάφους. Δεν υπάρχει πια αξιοπιστία όχι μόνο ως προς τις χώρες ΑΣΕΑΝ που ε, λαμβάνουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αν αγνοήσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες μέσω της ΕΙΕΔ να προωθήσουμε την καταπολέμηση των διακινητών. Ευχαριστούμε. Εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Ταραμπελαγιά, 1,5 λεπτό. Εάν η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία μεγάλη κρίση με μεγάλες ροές μεταναστών στη Μεσόγειο, θα πρέπει να στραφούμε προς την Νοτιοανατολική ε, Ασία επίσης. Επειδή είμαι αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, με τις χώρες ΑΣΕΑΝ, θα ήθελα να πω ότι οι Ροχίνια ζούσαν στη Βυρμανία και ζουν, αλλά είναι απάτριδες γιατί δεν τους χορηγείται η ηθαγένεια. Και μετά τις διώξεις τι κάνουν, διαφεύγουν προς την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία. Οι διακινητές βεβαίως χωρίς δισταγμό τους ε, οδηγούν σε μία νέα γη, άγνωστη γη. Και βλέπουμε ότι μετά την ε, ανακάλυψη των ομαδικών τάφων θα πρέπει να δράσουμε τάχιστα για να σταματήσουμε αυτή τη μεταναστευτική ροή που οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους προς το θάνατο. Οι Ροχίνγκια θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους Βιρμανούς. Χαιρόμαστε για την απόφαση της Μαλαισίας και της Ινδονησίας να θέσει τέρμα σε αυτή τη δίωξη και να υποδεχτεί χιλιάδες Ροχίνγκια μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης σε αυτό το μέρος του κόσμου, στην Νοτιοανατολική Ασία. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, του ECR, Μπασίρ, για ένα λεπτό. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες για τη βοήθεια τους έτσι ώστε να γνωστοποιηθεί το θέμα των Ροχίνια. Παρόλο που είναι πολύ αργά θα πρέπει να στυλιτεύσουμε τις κυβερνήσεις οι οποίες είναι άμεσα ή έμεσα υπεύθυνες για την ε, κατάσταση. Βλέπουμε ότι το Μιανμάρ έχει το, το χειρότερο γνώμονα για την δίωξη των ανθρώπων και θα πρέπει να, ε, ληφθεί, να αναλυφθεί η δράση έτσι ώστε να στυλιτεύσουμε την Μιανμάρ και να βγει αυτό το έθνος από το Μεσαίωνα και να βρεθεί στον 21ο αιώνα θα πρέπει να έχουμε μια κοινή κατανόηση. Φέρουμε ηθική ευθύνη όσον αφορά τη διάσωση ανθρωπίνων ζώων. Οι γείτονε ε, του Μιανμάρ δεν θα πρέπει να εργούν, θα πρέπει να διασώσουν τους Ροχίνια με βάση το δίκαιο της θαλάσσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Φιλελευθέρ, ο κύριος Ντεπρέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Όποιοι είδαν ε, το ρεπορτάζ ε, για την κατάσταση και για τα θύματα Ροχίνγκια, άνθρωποι που καίγονται ζωντανοί, ε, βιασμοί, αποκεφαλισμοί. Και όχι μόνο δεν γίνεται τίποτα στη χώρα για να τους προστατεύσουν, αλλά τους καταδιώκουν, να τους θερούν την θα τους. Όσοι βλέπουν και γνωρίζουν όλα αυτά, ξέρουν ότι και ο πρώτος υπεύθυνο για το Γολγοθά είναι η Βυρμανία και θα πρέπει πραγματικά να ανακαλέσουμε τη χώρα αυτή στην τάξη και να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να σεβαστεί ε, τη δήλωση για, τα, για την προσοχή των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε θα πρέπει να πάψει επίση ο αποκλεισμό τη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων ε, στου καταβλισμούς των προσφύγων Ροχίνγκια ε, στο Έδαφο τη Βερμανίας. Και τέλο, κύριε Επίτροπε, αν έχετε την καλοσύνη να με ακούσετε, έχω ένα ερώτημα. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, μου δίνετε τη δυνατότητα να σα κάνω μια ερώτηση παρακαλώ. Μου δίνετε τη δυνατότητα να σα κάνω μια ερώτηση για του Ροχίνγκια. Το 2012 αποφασίσαμε τη Βυρμανία να την επανετάξουμε στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Έτσι μπορεί να εξάγει τα προϊόντα της ε, χωρίς δασμούς, ε, ούτε ποσοστώσεις ε, στις ευρωπαϊκές αγορές. Μόνο τα όπλα και τα πυρομαχικά εξαιρούνται. Εάν η Βυρμανία συνεχίσει να παραβιάζει τόσο συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόθεση να θέσει υπό αμφισβήτηση αυτήν την επανένταξη στο σύστημα γενικών Τιμήσεων. Ευχαριστώ. εκ Πρασίνων Τζιν Λάμπερτ. λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω επισκεφθεί ορισμένου από του καταβλισμού ε, πληθυσμού Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντέ. Οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν ε, εδώ και δεκαετίες ε, να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή εκεί. Γιατί αυτά που βλέπουμε από τη Βερμανία και το Μιανμάρ είπαν πολύ ότι πρόκειται για μια πραγματική εθνοκάθαρση. Βλέπουμε ροχίνγκια που για γενιές ζούσαν εκεί ε, να χειραγωγούνται από την κυβέρνηση, να τους επιτρέπουν ε, να ψηφίζουν όταν συμφέρει την κυβέρνηση σε ψευτοεκλογές, ενώ τώρα αυτές τις λευκές κάρτες που είχα στη διάθεσή τους να τους τις στερούν τώρα, που δεν τους συμφέρει να ψηφίζουν. Ο λαός των Ροχίνγκια χρειάζεται άδεια από το κράτος για να συνάψει γάμο, για να αποκτήσει παιδιά. Δεν μπορούν να τους προστατεύσουν από την ε, φιλετική βία και από την κρατική βία και τους διωγμούς. Επομένως ε, δεν εκπλήσει το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς έχουν διαφύγει από τη χώρα. Και πάλι όμως ε, κινδυνεύουν και ε, να χειραγωγηθούν. Είναι σαφές, το είπαν και άλλοι, ότι η πηγή του προβλήματος είναι η Βερμανία Ανμάρ που ούτε καν δεν πήραν πίσω τα 200 και 300 άτομα που αναγνώρισαν ότι είναι πολίτες της χώρας. Ε, δεν τους έχω πάρει λοιπόν από αυτούς τους καταβλισμούς στο Μπαγκλαντές. Θέλω λοιπόν να προσθέσω τη δική μου φωνή και τη φωνή της ομάδας μου σε όσους λένε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα ε, απέναντι στην Περμανική κυβέρνηση για να ανταποκριθεί στις ευθύνε της και για να υποδεχθεί, να φροντίσει, να δώσει και ηθαγένεια στα άτομα αυτά που διώκει εδώ και τόσο καιρό. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πόσπισιλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταδικάσει τη βία κατά του λαού των Ροχίνγκια. Θα πρέπει να το κάνουμε και επίσημα. Αν η Βυρμανία δεν αλλάξει την πολιτική της, ε, αυτό θα πρέπει να έχει επιπτώσει στις αμοιβαίε σχέσεις μας και ε, η οικονομική επίπτωση, οι οικονομικές επιπτώσεις κατά της Βυρμανίας, γιατί ε, εκείνη είναι η υπέτεια για την παρούσα κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί η Ροχίνια έπρεπε να... δεν διαθέτουν πλέον ηθαγένεια. Γιατί τους αποσπάστηκε αυτό το δικαίωμα. Η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία, εάν δεν τηρήσουν το διεθνές δίκαιο, εάν δεν ρίξουν φως αυτά τα μεγάλα εγκλήματα, αυτό θα πρέπει να έχει επιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπετίνη έχει το λόγο. Πρόεδρε, βλέπουμε με το ψήφισμα το δράμα που σούν οι Ροχίνγκια που ε, διώκονται στις γείτονες χώρες. Κανένας δεν τους θέλει, διώκονται και βασανίζονται. Είναι απάτριδες. Δεν είναι άνθρωποι, αλλά φαντάσματα. Η Ευρώπη θα πρέπει να θέσει τις χώρες αυτές στη, υπό τις ευθύνες τους, αλλά εάν αυτό το δράμα των σκαφών που διαπλέουν τις θάλασσες δεν λυθεί, δεν θα λύσουμε ούτε το θέμα της ε, Μεσογείου. Σήμερα η Μαλαισία και η Ινδονησία αποφάσισαν να υποδεχτούν τους απελπισμένους. Όμως τα ευρωπαϊκά κράτη ε, σε σχέση με αυτό το καθεστώς ποσοστώσεων θα είναι εξίσου διατεθειμένοι να κάνουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο Ντάν Πρέντα έχει το λόγο μετά την ανακάλυψη των μαζικών τάφων στο Μιανμάρ και στη Ταϊλάδη βλέπουμε ότι πολλοί μετανάστες βρίσκονται στα χέρια των διακινητών. Υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί με την κρίση που ζούμε εμείς στο, στη Μεσόγειο. Είτε πρόκειται για την Νοτιοανατολική Ασία, είτε για τη Μεσόγειο, θα πρέπει να δοθεί μια λύση περιφερειακού χαρακτήρα και θα πρέπει στη διάσκεψη του Μπαγκόκ να δοθεί μια λύση. Δεν μπορούμε να παραπέμπουμε το θέμα στις ε, καλένδες όπως κάνει η Βυρμανία. Η χτεσινή συμφωνία μεταξύ Ινδονησίας, ε, Μαλαισίας και Ταϊλάνδης είναι κάτι το πολύ ε, θετικό, αλλά θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα της ηθαγένειας στους Ροχίνγκια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, είχε ζητηθεί αυτή η συζήτηση να γίνει το απόγευμα. Μετά μετατέθηκε το πρωί. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε περισσότερο κόσμο το απόγευμα παρά το πρωί όπως δείχνει η παρουσία εδώ των μελών. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Πέτχυρ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάνω από 140.000 πρόσφυγες Ροχίνγκα έχουν επιβιβαστεί σε σκάφη και σκαφίδια προκειμένου να διασωθούν. Είδαμε ότι πολλοί έχασαν το τελευταίο διάστημα τη ζωή τους προσπαθώντα να γλιτώσουν από το κατασταλτικό Καθεστώ. Καλωσορίζω λοιπόν τι αποφάσει τη Ινδονησία και τη Μαλαισίας να προσφέρουν άσυλο στους ανθρώπους αυτούς. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την ουσία του προβλήματος που είναι η πολιτική της Μιανμάρ. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να σταματήσουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εκμετάλλευση των Ροχίνγκια. Πρέπει να είναι ενιαία η αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σταματήσουν οι μαζικοί τάφοι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριος Φουζούλιντσα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, όλοι ξέρουμε ότι η Ροχίνγκια είναι η πλέον διοκόμενη εθνότητα στον κόσμο. Ε, γίνεται λαθρεμπόριο μέσω της Ταϊλάνδης και άλλων, περιοχών, και άλλων χωρών της περιοχής από δουλοεμπόρους που τους κρατούν σε στρατόπεδα αναγκαστικά εργασία, εργασίας, τους κρατούν όμοιρους, ε, τους ε, υποσυτίζουν μέχρι θανάτου. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και καλό τη Μιανμάρ να χορηγήσει ε, καθεστώς ισότιμου πολίτη και η ηθαγένεια πλήρη στους Ροχίνγκια για να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι απαράδεκτο επίσης το να ε, αποθούνται προς τη θάλασσα. Πρόκειται για παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και πρέπει αυτό να συζητηθεί στις επόμενες συναντήσεις με την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία και τη Μαλαισία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Νότη Μαριάς κύριε πρόεδρε η ανακάλυψη μαζικών τάφων με πρόσφυγες ροχίνγκια στη νότια ταϊλάνδη έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη. η περιοχή αυτή είναι το σταυροδρόμι του εμπορίου ανθρώπων και των δουλεμπόρων που οδηγούν τους πρόσφυγες σε φυλακές στρατόπεδα όπου επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες. Η ροχίνγκια είναι μια εθνοτική μειονότητα μουσουλμανικού θρησκεύματος η οποία καταπιέζεται από το βουδιστικό κράτος της μιανμάρ όπου η κυβέρνηση υπό τον έλεγχο του στρατού καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. για άλλη μια φορά χάνονται ζωές για θρησκευτικούς λόγους. εδώ τα θύματα είναι μουσουλμάνοι. σε άλλες περιοχές οι τζιχαντιστές είναι οι θύτες. όμως όπως έχουμε επισημάνει ξανά τα αίτια της φτώχειας και της ανέχειας δεν είναι θρησκευτικά ή εθνοτικά. οφείλονται στην οικονομική εκμετάλλευση των λαών από τις μεγάλες διεθνείς πολυεθνικές επιχειρήσεις. άμεση λοιπόν διακοπή διαπραγματεύσεων της ευρωπαϊκής ένωσης με την ταϊλάνδη προκειμένου να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει το ανθρώπινο εμπόριο να ληφθούν μέτρα στην περιοχή γιατί και στην ασία μπορεί να έχουμε μια νέα λαμπεντούζα. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ Ιάκοφτσιτς. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει με μια πολιτική απερίφραστη έναντι της Ασίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα δεινά δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, μαζικού τάφους, φρικαλαιότητες. Μιλάμε για απόπειρες ακόμη και εθνοτικής κάθαρσης. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις έναντι της Ινδονησίας, έναντι της Μαλαισίας, αλλά κάποιες προθέσεις πρέπει να τις αναθεωρήσουμε και αυτές αφορούν τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη. Πρέπει να πούμε στις χώρες αυτές ότι ναι, είμαστε στο πλευρό σας, ναι, είμαστε φίλοι σας, αλλά πρέπει και εσείς να κάνετε ό,τι οφείλετε για το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ευχαριστώ κύριο Καστάλντο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μου φαίνεται φοβερή αυτή η κατάσταση. Θεωρείται ότι η Ροχίνια είναι ο λαός που διώκεται περισσότερο ανά τον κόσμο. Από το 82 και μετά δεν μπορούν στη Βυρμανία ούτε να έχουν την ηθαγένεια, ούτε να την αποκτήσουν και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν περισσότερο από δύο παιδιά. Αυτό αποτελεί κατάφορη, κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι ενός λαού. Δυστυχώς πρέπει να καταφύγουν σε όμορες χώρες και βεβαίως εκεί προωθείται το δουλεμπόριο, οι διώξεις και ε, δυστυχώς ε, υπάρχουν καταστάσεις που θυμίζουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του ναζισμού. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει βία, διακρίσεις, ρατσισμός και έλλειψη τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν συνεχίσουμε να έχουμε εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές, η κατάσταση αυτή δεν θα επιληθεί. Ας είμαστε υπεύθυνοι για μια φορά. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια είναι ιδιαίτερα αδεινή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την ανθρωπιστική κρίση βλέποντας ε, το ότι οι Ροχίνγκια πρέπει να καταφύγουν στο ε, Μπαγκλαντές και δυστυχώς ε, τα σκάφη αυτά διαπλέουν τις θάλασσες χωρίς να φτάσουν πουθενά. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις αυτά τα κράτη καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα η προτεραιότητα είναι να σώσουμε ζωές και όχι να ε, τις θέσουμε, να θέσουμε περισσότερο ζωές σε κίνδυνο. Αυτό είναι, πιστεύω, και, το, και η έκβαση της διάσκεψης μεταξύ των τριών χωρών ε, Ταϊλάνδης, ε, Μαλαισίας και Ινδονησίας και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον θα δοθεί προσωρινό άσυλο σε αυτούς τους ανθρώπους που τους έφερε η θάλασσα. Παράλληλα θα γίνει μια περιφερειακή διάσκεψη στην Ταϊλάνδη στις 29 Μαΐου για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, διότι χρειάζεται περιφερειακή απάντηση για να μπορέσουμε να στυλιτεύσουμε το διασυνοριακό ε, έγκλημα και για να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της κακοδαιμονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την ΑΖΕΑΝ να αντιμετωπίσει δραστικά το ζήτημα, να αναλάβει ενεργό ρόλο και βεβαίως αυτό που έχει σημασία πρωτίστως είναι η ευημερία των ε, μειονοτήτων, της μειονότητας των Ροχίνγκια στο Μιανμάρ, που είναι η χώρα από την οποία προέρχονται οι περισσότεροι Ροχίνγκια. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει δραστικά το ζήτημα η κυβέρνηση του Μιανμάρ και θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μόνο αν αναγνωριστούν οι Ροχίνγκια θα δοθεί τέλος σε αυτή τη μαζική έξοδο των Ροχίνγκια. Ροή η οποία έχει αυξηθεί δραματικά πρόσφατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην εμπροστοφυλακή για ε, βιώσιμες λύσεις για τους Ροχίνγκια. Η κατάσταση μας απασχόλησε τα τελευταία χρόνια στον πολιτικό διάλογο με το Μιανμάρ ιδιαίτερα στον ε, διάλογο του επίπεδου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποβάλλουμε ψηφίσματα και προτάσεις στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να αναγνωριστεί η κατάσταση αυτή που επικρατεί στο Μιανμάρ. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και αναπτυξιακή αναγνωρίζοντας το καθεστώς αυτό ε, στο Μιαν, του Μιανμάρ. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διώκονται πια οι Ροχίνγκια και να μην χρειάζεται να καταφεύγουν στο Μπαγκλαντές. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη των, ε, μαζικών, των ομαδικών τάφων στη Νότια Ταϊλάνδη και μετά από την ανακάλυψη των στρατοπέδων κράτησης. Οι, άνθρωποι, οι ανθρώπινες ζωές δεν είναι αγαθά. Δεν είναι εμπόρευμα. Ζητήσαμε από την Ταϊλάνδη να καταπολεμήσει την διακίνηση των ανθρώπων καθώς και την αναγκαστική εργασία στα σκάφη και στα αλλιευτικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα συμπράξει με τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ για την συζήτηση και για το ψήφισμα αυτό το οποίο μιλάει από μόνο του. Έχω καταγράψει όλα σας τα σχόλια, θα τα συζητήσω με την Αντιπρόεδρο Φεντερίκα Μογκερίνη. και θα προσπαθήσουμε η δράση μας να είναι πιο αποτελεσματική. γιατί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ενεργοί και δραστικοί στην αντιμετώπιση του θέματος των προσφύγων Ροχίνγκια. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφίσματος, λίγη η συζήτηση και η υπάρχει και μια πρόταση από το EFFD, τους πράσινους, τους φιλελεύθερους, το ECR, e, την ΚΟΕ, e, καθώς και τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Λίγη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αμέσως μετά τη συζήτηση, την επόμενη συζήτηση, δηλαδή στις 12. Περνάμε στην επόμενη συζήτηση.